So, good afternoon. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων, αγαπητοί καλεσμένοι, έχω τη χαρά να σας καλωσορίσω σήμερα το απόγευμα στο εργαστήριο Παριθμών 5 σε σχέση με την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, στο οποίο, στην οποία επιτροπή είμαι και εγώ, και επίσης και από την οργάνωση UN Women. Θα δούμε τους ε, στόχους ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και θα εστιάσουμε περισσότερο στην ισότητα των φύλων, στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για την αξιοπρεπή εργασία για να δούμε πώς αυτοί οι στόχοι βοηθούν την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Η συζήτηση αυτή θα αντιμετωπίσει τις συστάσεις του υψηλού επίπεδου πάνελ του ΟΗΕ για τα θέματα των γυναικών και τον οδικό χάρτη του UN Women για την ουσιαστική ισότητα δρόκη και γυναικών το 2030. Ο στόχος του εργαστηρίου λοιπόν είναι να ταυτοποιήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο εμείς ως μέλη του Κοινοβουλίου σε όλα τα μέρη του κόσμου μπορούμε και θα πρέπει να διαδραματίσουμε ένα ρόλο στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απόλυτα προσιλωμένο στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Στις πρόσφατες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14 Φεβρουαρίου 2017 προς το Συμβούλιο για τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την ε, επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για το καθεστώς των γυναικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ιδίως ο στόχος υπεριθμών 5 αποτελούν την επίτευξη ισότητος ανδρών και γυναικών και τη χειραφέτηση των κορισιών και των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλο το θεματολόγιο του 2030 και στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η χειραφέτηση των γυναικών λοιπόν σημαίνει να τους δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνουν ανεξαρτητά, οικονομικά ανεξάρτητες, να έχουν ίση εκπροσώπηση σε όλη την κοινωνία μας, να διαδραματίζουν ίσο ρόλο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και να έχουν περισσότερη παρουσία στη δημόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Συγχρόνως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι μία από τις προτεραιότητες μας θα πρέπει να είναι να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες να υποστηρίζουν την αξιοπρεπή εργασία και την απασχόληση για όλες τις γυναίκες. Πριν ξεκινάσουμε το έργο μας, θέλω να σας υπενθυμίσω κάποιες διαδικαστικές πλευρές. Η για αυτό το εργαστήριο θα είναι η κυρία Τζάνσον. Θέλω να την ευχαριστήσω για το έργο το οποίο έχει αναλάβει. Θα προετοιμάσει μια έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει και τα συμπεράσματα του εργαστηρίου μας και αυτά τα σχόλια θα παρουσιαστούν, αυτά τα συμπεράσματα συγγνώμη, θα παρουσιαστούν αύριο το πρωί. Θα ήθελα τώρα για τη συζήτηση, θα ήθελα να ζητήσω από όλους και όλες εσάς που θέλετε να λάβετε το λόγο, να δώσετε στους κλητήρες το όνομά σας και το φορέα από τον οποίο προέρχεστε, το Κοινοβούλιο, για να λάβετε το λόγο οι Πρέπει να γίνει αυτό μέσα στα επόμενα 15 λεπτά. Αν υπάρχουν πολλές αιτήσει, θα πρέπει να κλείσω ο κατάλογος Και τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω τους ομιλητέ μας. Πρώτα απ' όλα την κυρία Αλία Ελ Γιασίρ, που είναι αναπληρώτρια του UN Women για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ για την παρουσία σας και επίσης τον κύριο Αυγούστο Λόπε Κλάρος, ο οποίος είναι ο διευθυντής του, της ομάδος παγκοσμίων δικτών για την ε, ε, ανάπτυξη στην ε, Παγκόσμια Τράπεζα στη Ουάσιγκτον. Πρώτα απ' όλα λοιπόν δίνω το λόγο στην κυρία Αλή Ελγιάσερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για αυτό το κομμάτι της εργασίας. Νομίζω πριν μίλησα για τους ε, στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, όμως ε, θα ήθελα πριν προχωρήσω να σημειώσω ότι πριν από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης είχαμε μια σειρά οκτώ στόχων που ήταν γνωστοί ως στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη, που υιοθέτησε η Εθνής Κοινότητα το 2000 και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, ε, υλοποιηθεί έως το 2015 υποτίθεται πως θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί στο 2015. Ωστόσο, οι ε, στόχοι της χιλιετίας είναι διαφορετικοί από αυτούς της βιώσιμης ανάπτυξης. Απαιτούνται δηλαδή διαφορετικά πράγματα. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης αφορούσαν μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι στόχοι της ε, βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν όλες τις χώρες. Ε, ένα γενικότερο θεματολόγιο λοιπόν. Και έτσι και τι είχαν αυτόνομο στόχο την ισότητα των φύλων και οι δύο κατηγορίες στόχων εδώ με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης χρειάζεται πιο σοβαρή και μόνιμη στράτευση και προσήλωση για την ισότητα των φύλων και αυτό όχι μόνο μέσω του αυτόνομου στόχου, του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθμών 5, αλλά πρέπει σε όλους τους άλλους στόχους εγκάρσια να εφαρμόζονται πολιτικές με στόχο την ισότητα των φύλων. Επομένως το 50-50 που λέμε έως το 2030 για ολόκληρο τον πλανήτη ως ισότητα των φύλων είναι στόχος ο οποίος εγγράφεται, ενσωματώνεται σε όλους τους στόχους της βιώσιμης, της ανάπτυξης. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε λοιπόν φέτος ε, τις γυναίκες σε ένα μεταλλασσόμενο χώρο εργασία ή κόσμο εργασία. Είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει και στην Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών CSW στις, ε, στη Νέα Υόρκη από τις 13 έως τις 24 Μαρτίου. Δηλαδή ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα. Αν την έκθεση ε, του του επίπεδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο Leave no one behind, μην αφήσετε κανένα πίσω. Ε, επτά μοχλοί τη ε, ε χειραφέτηση των γυναικών, οικονομική χειραφέτηση έχουν καταγραφεί. Βεβαίω δεν θα μπω στι λεπτομέρειε, μπορείτε να του δείτε όλου ε, στη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και οφείλουμε να συζητήσουμε υπόψη όλων αυτών των μοχλών Τη ε, οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν συγκεκριμένα το έργο αυτή τη ε, ομάδα εργασία του workshop. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω κάποια από τη δουλειά που κάνουμε εμεί ω γυναίκε εν του στόχου υπαριθμών 5, ε, αλλά και του υπαριθμών 1 για την αντιμετώπιση τη φτώχεια με κάθε τη μορφή παντού, του 8 για την βιώσιμη παραγωγική και ανοιχτή ανάπτυξη, απασχόληση, αξιοπρέπεια στην απασχόληση για τους πάντες και υπαριθμών 10 για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ όλων και μεταξύ των κρατών. Και ιδιαίτερα οι δύο μοχλοί που υπογράμμισε το πάνελ υψηλού επίπεδου αφορούν πρώτον την νομική υποστήριξη και τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας όταν αυτή επιβάλλει διακρίσεις και δεύτερον αναγνώριση, ε, περιορισμός και ανακατονομή της αμοιβή και της εργασίας αυτή αμοιβόμενη ήμη. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τον υπαριθμό 1, κατάργηση κάθε, 5, ε, κατάργηση κάθε διάκριση βάρος των γυναικών. Στο 5.1.1 επικεντρωνόμαστε στο κατά πόσο υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την προαγωγή, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της αποτροπής των διακρίσεων που θα στηρίζονταν ενδεχομένω στο φύλλο. Θεωρούμε ότι αυτός ο δείκτης θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για την παρακολούθηση αλλά και για την επιτάχυνση των προγραμμάτων. Ως ε, γυναίκες λοιπόν εργαζόμαστε στη μεθοδολογική ανάπτυξη των δικτών αυτών σε συνεργασία με, την, ε, με τις ομάδες εργασίας. Ιδιαίτερα έχουμε ένα εργαστήριο πέρσι τον Ιούνιο ε, που επεξεργάζεται αυτόν τον δίκτυ και ιδιαίτερα την αντίληψη ε, και σχεδιασμό του, αλλά και τις πηγές του δικαίου που θα πρέπει να εξετάζονται. Συλλογή λοιπόν δεδομένων ε, από διάφορες έρευνες και χώρες ε, διαφόρων περιοχών του κόσμου που κλήθησαν να συνεργαστούν για τη συλλογή αυτών των δεδομένων και όπως υπόθηκε και νωρίτερα μέσα στο πλαίσιο πάντα της, του στόχου ε, για το 2030 έχει χαραχθεί ο στόχος ε, για το 2030 για τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις, κυβερνήσεις, ε, κοινοβούλια, κοινωνία, με στόχο δηλαδή την κατάργηση, εξάλληψη, μεταρρύθμιση νομοθεσίας που έχουν να κάνουν ε, με ζητήματα ισότητας των φύλων και διεθνού προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ σε ένα άλλο καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε η, ομάδα, η Επιτροπή των Γυναικών των Εθνών, ειδικά στα Βαλκάνια, με στόχο την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης θέσης του φύλου σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το κεκτημένο για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπληρώνει κάθε στόχο και την υλοποίηση ε, μέτρων για την αηφόρο ανάπτυξη προς όφελος γυναικών αλλά και ανδρών και αγοριών, ε, όπως και κορίτσιων φυσικά. Ιδιαίτερα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τη βία ει βάρο των γυναικών. Χώρε τη Νοτιοανατολική λοιπόν Ευρώπη μπορεί να επεξεργάζονται και να ε, προωθούν τι ε, διαδικασίε για την ένταξη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχύουν τα σώματα που προάγουν την ισότητα των φύλων και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω αυτού του μέσου ε, του facility για την ισότητα των φύλων. Βεβαίω δεν αρκεί να περνάνε νόμοι, πρέπει και να εφαρμόζονται και να ελέγχεται η επιβολή τους. Ο κύριος Κλάρος, με τον οποίο είναι χαρά την τιμή να συνεργάζομαι, θα σας μιλήσει περισσότερο για τις λεπτομέρειες σχετικές με την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, επομένως προς τις λεπτομέρειες σας τις δώσει εκείνος. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι ελπίζουμε πως οι ε, πρωτοβουλίες αυτές θα επιταχύνουν την πρόοδο της δουλειά μας στον τομέα αυτό και έτσι θα έχουμε έως το 2030 εγγύξει το στόχο ώστε καμία χώρα να μην έχει νομοθεσία ενισχύ εις βάρος των γυναικών που θα διακρίνει δηλαδή ει βάρος των γυναικών. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και ενσωμάτωση και άνοιγμα των θέσεων, τη θέσης της γυναίκας στην οικονομική ζωή. Αυτό σημαίνει και θεσμική φραγμή, όπως ε, δημοσιονομικά, όπως δυσκολίε, άλλε οικονομικές να ε, εξαλειφθούν, ώστε να είναι ανοιχτέ οι δυνατότητε για ομάδες ανθρώπων εν γέννη, ανδρών, γυναικών, παιδιών, ε, είτε αγοριών είτε κοριτσιών. Ε, για οικονομική ανάπτυξη. Το κόστος για την παγκόσμια οικονομία, όπως άλλως αναφέρθηκα και νωρίτερα, από, τις, ε, από τη διακριτική θεσμική μεταχείριση, αλλά και τη βία εις βάρος των γυναικών, ξεπερνά τα 11 τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και πρέπει να κοιτάξουμε τις περιφερειακές παρεμβάσεις για την ε, τα τις, γλω... τις γνώσεις της ε, τεχνογνωσίας ε, σε όλο τον κόσμο και αυτό βέβαια ξεκινώντας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. Επί παραδείγματι, ύστερα από πέντε χρόνια επενδύσεων της, Επι... Ε, Επιτροπής για τις Γυναίκες σε θετικές ως προς την ισότητα των φύλων δραστηριότητες δημοσιονομικές στην Αλβανία, 61 εκατομμύρια ευρώ έχουν αποδεσμευτεί σε εθνική χρηματοδότηση και το 2017 αναμένεται ότι 11 υπουργεία Τη Αλβανία θα έχουν δεσμεύσει 85 εκατομμύρια ευρώ για θέματα γυναικών ή ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερα λοιπόν ε, σημασία έχει αυτό να κοιτούμε ε, το, το ζήτημα της αποδέσμευσης, τη της ε, απαλλαγής από την ε, κρατούμενη προσέγγιση των προϋπολογισμών και σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Ε, υπάρχουν παρεμβάσεις από την Επιτροπή των ΗΠΑ για τις γυναίκες, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολλά θέματα, αλλά ξεκινούμε με ένα παράδειγμα από έναν και μόνο Δήμο, με την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, παραδείγματι, που σήμαινε πρόσβαση για 15.000 γυναίκες της υπαίθρου. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Έχουμε προσεγγίσεις ε, κατά των διακρίσεων, ανεξαρτήτως ε, κοινωνικο-οικονομικού καθεστώτος, αναπηρίας, ενδεχόμενης γεωγραφικής θέσεως, εθνότητας και συναφών διακρίσεων. Κανεί δεν πρέπει να μείνει πίσω. Αυτό είναι το συνθημά μα και ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε τον όρο της εργασίας και της κατανομής της εργασίας. Αυτό ιδιαίτερα το υπογραμμίζει το πάνελ υψηλού επίπεδου του ε, ε, Γενικού Γραμματέα. Ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης παριθμών 5 ορίζει 9 στόχους, 9 στοχεύσεις, ιδιαίτερα ε, για την αναγνώριση και την αξιοποίηση λόγηση, την πρόσδοση αξίας δηλαδή στην δουλειά και την μέρημνα τη φροντίδα που προσφέρουν οι γυναίκες στο σπίτι μέσω από την εξασφάλιση δημοσίων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας και προαγωγής κοινή ευθύνη. Πρέπει να αναγνωριστεί λοιπόν αυτό, γιατί άλλωστε η μη αμοιβόμενη εργασία των γυναικών υπήρξε ένα από τα κύρια εμπόδια στην ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας και λειτουργεί εις βάρος και της απασχόλησης. Έχουμε δυόμιση φορές περισσότερες ε, απλήρωτες γυναίκες στην Αλβανία 77% των γυναικών δουλεύουν περισσότερες ώρες στην Αλβανία, 55% στην ε, Τουρκία. Σε περιοχές της Ευρώπης Κεντρικής Ασίας, ε, στο χώρο της φροντίδας των φροντιστών, που έχει πάρει πολύ μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει μία αμοιβόμενος ε, χώρος εργασίας, μία αμοιβόμενη απασχόληση, βλέπουμε ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας και οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών. Χρειάζονται λοιπόν υποδομές και κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας, υπηρεσίες, υπηρεσίες για τα παιδιά, τον ασθενή, τον ηλικιωμένο, το άτομο με αναπηρία, που μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη και πάλι μέσα σε ένα πλαίσιο λιτότητας και ύφεσης. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή έτσι να δημιουργήσουμε απασχόληση για άντρε και γυναίκε και να προαγάγουμε μια ανοιχτή προ όλου ανάπτυξη για την ισότητα των φύλων, για την ενίσχυση του οικονομικού περιβάλλοντο. Η, η παροχή κοινωνικής λοιπόν μέρημνας ε, είναι μια λύση την οποία ελπίζουν περισσότερες χώρες θα υιοθετήσουν για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ έχουμε να κάνουμε και μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που δίνουν και οικονομική χειραφέτηση στις γυναίκες αλλά και οικονομική πολιτική για όλες τις χώρες. Η χειραφέτηση λοιπόν των γυναικών θα καλυφθεί σε μια δεύτερη έκθεση στην προσεχή σύνοδο τη Επιτροπής για το καθεστώ των γυναικών μεταξύ των διαφόρων διαβουλεύσεων που έγιναν για την πρώτη και τη δεύτερη έκθεση συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών διαβουλεύσεων που έγιναν εδώ στις Βρυξέλλες εξασφαλίστηκε ευρύτερη συνένεση ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές δεν έχουν ουδετερότητα, δεν είναι ουδέτερες απέναντι στο φύλλον και χρειάζονται υπεύθυνε οικονομικές πολιτικές ιδιαίτερως, αλλά και μακροοικονομικές πολιτικές ε, ακόμη περισσότερο. Εμείς ελπίζουμε από τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα βοηθήσουμε με μια εκτεταμένη ε, έκθεση που θα καλύπτει την θέση των γυναικών και στο εμπόριο και την ανάπτυξη, ώστε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της ε, κοινωνικο-οικονομικής ε, πολιτικής. Μπορεί να σας φαίνεται τεχνοκρατικό αυτό, αλλά μια χρηματοδότηση και οικονομικές δημοσιονομικέ πολιτικέ που θα λαμβάνουν υπόψη την διάσταση του φύλου, θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην α, χειραφέτηση στην οικονομική των γυναικών. Εδώ μπορεί να έχουμε ένα τεράστιο βήμα μπρο για την ισότητα των φύλων χάρη σε τέτοιου πολιτικέ και τα κοινοβούλια έχουν τεράστιο ρόλο να διαδραματίσουν προ την κατεύθυνση αυτή. Με βάση μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο οι βελτιώσει ω προ την ισότητα των φύλων θα οδηγούσαν σε 10,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας περισσότερες έως το 2050. Ε, γι' αυτό λοιπόν το ποσοστό απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το 80% και το ΑΕΠ κατά κεφαλήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει θετική εξέλιξη με αύξηση μέχρι και 10% έως το 2050. Όταν λοιπόν αναζητούμε συγκεκριμένε λύσει και θέλουμε να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την οικονομική χειραφέτηση τη γυναίκα, λύσει έχουμε στη θέση μα. Έχουμε όμω ακόμα 13 μόλις χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανισότητας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης το 2030. Χρειάζονται λοιπόν οικονομικές ε, ε, και εταιρικές σχέσεις για να βοηθήσουμε όλοι να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αλιασίρ για την παρέμβασή σας και τώρα δίνω το λίγο στον κύριο Λόπες Κλάδος. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι, με μεγάλη χαρά που μπορώ να είμαι μαζί σας για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Στην Παγκόσμια Τράπεζα. Εδώ και κάποια χρόνια έχουμε πολλά σχετικά προγράμματα. Εξετάζουμε το δίκαιο σε 173 χώρες και κοιτάζουμε πώς χρησιμοποιεί την νομοθεσία για να γίνεται διάκριση κατά των γυναικών. Κοιτάζουμε το σύνταγμα, το οικογενειακό δίκαιο, το εργασιακό, μια σειρά από νομικά μέτρα και κοιτάζουμε τους νόμους για να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρξει διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών τρόπον τεινά, για να περιοριστούν οι ευκαιρίες που τους προσφέρονται. για να υποβαθμιστούν, για να μην μπορούν να συμβάλλουν πλήρως στην ε, παραγωγή πλούτου και την ευημερία, Βεβαίως, πριν από την ίδρυση αυτού του προγράμματος που ονομάζεται «Γυναίκες ε, επιχειρήσεις και νόμος», ξέραμε ήδη ότι σε κάποιες ε, χώρες το δίκαιο αποδίδει τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας στον σύζυγο. Δεν μπορεί δηλαδή μια γυναίκα να ιδρύσει μια επιχείρηση χρησιμοποιώντα ε, για να πάρει δάνειο μια υποθήκη του σπιτιού. Σε κάποιες χώρε ο νόμος ε, χρησιμοποιείται για να επιβληθούν περιορισμοί στις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων. Το ωράριο εργασία του. Επίση, είναι χαρακτηριστική η κλάδη στου οποίου απασχολούνται οι γυναίκε. Θα σα δώσω κάποια παραδείγματα ε, εντό ολίγου. Και αυτό εντείνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πριν από λίγα χρόνια, λοιπόν, αρχίσαμε να θέτουμε μια σειρά από ερωτήματα για τα οποία ψάξαμε τι απαντήσει στην νομοθεσία σε αυτέ τι 173 χώρε. Μπορεί μια γυναίκα να βρει δουλειά όπω ένα άντρα. Μπορεί να εγγράψει μια επιχείρηση όπως μπορεί να την εγγράψει ένας άντρας. Μπορεί να πάρει εθνική ταυτότητα. Μπορεί να ταξιδέψει με την ίδια ελευθερία όπως ένας άντρας. Έχει ίδια δικαιώματα ιδιοκτησίας. Επιβάλλονται περιορισμοί από τον νόμο για το τι δουλειά μπορεί να βρει, σε τι κλάδους μπορεί να απασχοληθεί. Υπάρχουν ποινικέ κυρώσει ε, για την σεξουαλική παρενόχληση την ενδοοικογενειακή βία. Είναι θεσμικό στο φύλλο προστατευόμενο. Και ούτω καθεξή. Δεν θα πω άλλα ερωτήματα. Απλώ φτιάξαμε αυτή τη τεράστια βάση δεδομένων και θα ήθελα να αξιοποιήσω τα λεπτά που μου διατίθενται για να σα παρουσιάσω μερικά τα πιο ενδιαφέροντα πορίσματα που προέκυψαν από, 100, από την έκθεση του 2016. Το πρώτο, στοιχείο είναι ότι μόνο σε 18 χώρες από 173 ο νόμος δεν επιβάλλει κανένα είδους περιορισμό. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι τυφλός ως προς το φύλλο. Δηλαδή, για να το θέσω διαφορετικά, σε 90% των χωρών υπάρχει τουλάχιστον ένα, για να μην πω 10, 25 περισσότεροι περιορισμοί, αλλά τουλάχιστον ένας αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι στι 18 αυτέ χώρε που δεν έχουν κανένα περιορισμό ω προ το φύλλο, η εικόνα είναι πολύ ανάμεικτη. Όντω, σε χώρε όπω η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Ισπανία, ο νόμο είναι εντελώ τυφλό, θεότυφλο ω προ το φύλλο. Μεταχειρίζεται ακριβώ με τον ίδιο τρόπο ε, άνδρες και γυναίκες. Όμως χώρες όπως η Δημοκρατία του Αγίου Δομήνικου, ή άλλες χώρες δεν ε, φαίνεται ξεκάθαρο για το εάν ο μισθό είναι ένα κριτήριο για να υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε 100 χρόνια για να υπάρξει μισθολογική ισότητα δηλαδή. Οι χώρες που είναι αναπτυγμένες με υψηλότερο εισόδημα έχουν δικαιότερη νομοθεσία προς τις γυναίκες υπολογίζοντας τον αριθμό των ε, περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος στις γυναίκες και υπάρχουν 30 χώρες στον κόσμο που υπάρχουν δεκάδες περιορισμοί και παραπάνω, όπως ε, οι περιοχές ε, της νότιας και της κεντρικής Αφρικής, μπορούμε να τα συσχετίσουμε με άλλα ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία. Αυτό που προκύπτει ως επισκόπηση είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσο πιο μεγαλύτερους περιορισμούς στον νόμο αντοπίσουμε σε μια χώρα, τόσο χαμηλότερη είναι η συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστά ως προς τους άντρες. Και είναι ε, λογικό αυτό. Οι περιορισμοί έχουν αποθαρρυντικό αποτέλεσμα στην διάθεση των γυναικών και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Και όσο περισσότεροι είναι οι περιορισμοί, τόσο λιγότερες γυναίκες ε, έχουν επιχειρήσεις. Όσο, περισσότερες είναι, όσο περισσότεροι είναι οι περιορισμοί, τόσο μεγαλύτερο είναι το μισθολογικό χάσμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο των περιορισμών, ε, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό των γυναικών που γράφονται στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με τα αγόρια μάλλον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν οι μητέρε ε, πιέζουν, ε, ή μάλλον δεν εργάζονται, τότε κάποια στιγμή τα παιδιά παρατάνε, τα κορίτσια παρατάνε το σχολείο. Ή αν εργάζονται, μάλλον παρατάνε πιο εύκολα το σχολείο για να καλύψουν κάποιε ανάγκε τη οικογένεια. Ε, κάποιε άλλε ιδέες πολλές χώρες σε πολλά μέρη του κόσμου επιβάλλουν έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό περιορισμό ε, για την απασχόληση. Τον περασμένο Απρίλιο πήγα στη Μόσχα, λιγότερο από χρόνο πριν, και ε, ε, συζήτησα με έναν υφυπουργό που ασχολείται με κάποια οικονομικά ζητήματα. Και προς το τέλος της συνεδρίασης γύρισα και μου είπε, κύριε Λόπες Κλάρος, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στη Ρωσία για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για την κοινότητα των επιχειρήσεων. Και μου ήρθε και του είπα, κοιτάξτε κύριε Υφυπουργέ, μήπως τις 456 δουλειές ε, που απαγορεύεται να πάρουν οι γυναίκες, να δουλέψουν οι γυναίκες στη Ρωσία, να τις καταργούσατε. Δηλαδή τις 456 περιορισμούς. Ε, και μάλιστα είχα μπροστά μου ένα κατάλογο με τι 456 αυτέ περιπτώσει και ήμουν έτοιμο και να τον βγάλω τον κατάλογο και να τι αναφέρω τι περιπτώσει αυτέ εφόσον χρειαζόταν. Αυτά υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα, την ε, ανάπτυξη, την πρόθεση των γυναικών ε, στην αγορά και δίνουν το μισθολογικό χάσμα προφανώ. Είναι πολλέ οι επιπτώσει για την οικονομική ε, ευημερία. Θα ξέρετε ότι πριν από λίγα χρόνια στα πλαίσια αυτού του προγράμματο αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία για την βία κατά των γυναικών και την σεξουαλική παρενόχληση. Η ερμηνεία από τα δεδομένα που προκύπτει από αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά ε, φοβερά εντυπωσιακή. Εάν κάνουμε σύγκριση με τον χωρών όπου υπήρξε νομοθεσία για την προστασία των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία και τις χώρες που δεν υπήρχε καμία τέτοια νομοθεσία όπω η Ρωσία, το Ιράν, η Αίγυπτος και άλλε πολλέ, προκύπτει ότι το μέσο, ο μέσος όρος προσδοκίμου των γυναικών είναι υψηλότερο, υψηλότερος εκεί όπου η νομοθεσία προστατεύει τις γυναίκες από τη βία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ως στοιχείο. Με άλλα λόγια, η νομοθεσία αυτή έτσι καλώς είναι πρόσφατο φαινόμενο. Εάν πάμε στην δεκαετία του 90, πριν από 25-26 χρόνια δηλαδή μόλις, μια χούφτα χώρε είχαν τέτοια νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία. Έκτοτε, ο αριθμό των χωρών έχει αυξηθεί. 127 χώρε έχουν τέτοια νομοθεσία. Στην τράπεζα, μαζί με άλλου συναδέλφου, έχουμε εκπονήσει μελέτη που κοιτάζει το θέμα τη πρώιμη θνησιμότητα των τελευταίων 50-60 ετών σε σχέση με την έλλειψη νομικής προστασίας για τις γυναίκες νομοθεσία που να προστατεύει από την ενδοοικογενειακή βία. Και τα στοιχεία που προκύπτουν είναι πραγματικά ε, καταθλιπτικά. Εκατομμύρια γυναίκες πέθαναν πρόεμα τα προηγούμενε δεκαετίες λόγω της έλλειψης προστασία τους. Σήμερα υπάρχει μια πολύ ζωντανή συζήτηση, καυτή συζήτηση για το όλο θέμα τη ανισότητα. Υπάρχει η εντύπωση ότι η ανισότητα είναι εκτό ελέγχου. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε στην Παγκόσμια Τράπεζα δείχνουν ότι οι ανισότητε μεταξύ των χωρών, οι ανισότητε εντό των χωρών μια ίδια χώρα, όπω και αν τα καταμετρήσουμε, δείχνουν ότι πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα θέλαμε. Δείχνουν ότι υπάρχει συγκέντρωση του πλούτου σε ένα πολύ στενό κύκλο αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι από τα στοιχεία για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις, όπου χώρες έχουν προβλέψει κίνητρα που διευκολύνουν τις γυναίκες να εργαστούν, όπως η άδεια για τους ε, πατέρες, ε, η ε, ε, απαγόρευση της απόλυσης μιας γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης, εκεί τα επίπεδα ανισότητα είναι χαμηλότερα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι μας λείπουν οι πολιτικές συστάσεις, γιατί το πρέπει να κάνει η νομοθεσία ε, για να καταπολεμήσει την ανισότητα. Είναι απλή απάντηση. Πρέπει να διευκολύνουμε τι γυναίκε να εργαστούν. Πρέπει να απαλληφθούν οι περιορισμοί. Αυτό θα έχει ένα πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην δυνατότητα των γυναικών να ενταχθούν στην εργασιακή δύναμη των διαφορών χωρών. Είναι πολλά τα αριθμητικά στοιχεία, δεν έχω χρόνο να σας τα αναλύσω σήμερα. Υπάρχει και άλλο ένα κριτήριο που θα μπορούσα να αναπτύξω, αλλά καλύτερα να ολοκληρώσω με μια-δυο παρατηρήσεις. Η ύπαρξη των δεδομένων ήδη οδηγούν σε σκέψεις και προκαλούν ένα κύμα μεταρρυθμίσεων από τον κόσμο. 95 μεταρρυθμίσεις είδαμε να ε, υλοποιούνται σε 64 χώρες πέρσι, όταν λέω ενώ εξαλείψεις συγκεκριμένων περιορισμών όπω του εντοπίσαμε εμεί στην έκθεσή μα. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Όλο και περισσότερε χώρε έρχονται στην Παγκόσμια Τράπεζα και λένε βοηθήστε μα. Βοηθήστε μα να αλλάξουμε την νομοθεσία μα ή τέλο πάντων έρχονται να μα πούν ότι άλλαξαν το, ε, τον αστικό κώδικα ή κάτι σε θεσμικό επίπεδο για να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, να απαλείψουν περισσότερες, περιορισμού. Αυτό είναι θετικό, είναι θετικές οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα και σιγά σιγά συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί νομικά ένα καλύτερο, ασφαλέστερο περιβάλλον. Με περισσότερη ισοτιμία για γυναίκες και άνδρες. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την ολόνα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι η ισότητα των φιλών ίσως να μην σημαίνει ή ότι μάλλον δεν είναι ένα παιχνίδι που ένας κερδίζει και άλλος χάνει. Δεν σημαίνει ότι οι άνδρες πρέπει να χάνουν όταν υπάρχει ισότητα. Σημαίνει ότι φτάσαμε σε ένα σημείο τη εξελικτική πορεία τη ανθρωπότητα που το να είναι κανεί αγόρι-κορίτσι δεν είναι καθοριστικό παράγοντα για το τι είδου ευκαιρίε θα να έχει στη ζωή του. Το τι επίπεδο πλούτου πρέπει να κατακτήσει. Να ολοκληρώσω λέγοντά σα κάτι που το βρίσκω μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Το φύλλο και την ισότητα τα βλέπουμε από μια ανθρώπινη σκοπιά προφανώς και στην Παγκόσμια Τράπεζα λέμε ότι η ανισότητα έχει και οικονομική επίπτωση. Προφανώς είναι κακό για την παραγωγικότητα, για την οικονομία, για την ε, ευημερία της ανθρωπότητας. Όμως η ανισότητα έχει και μια ηθική διάσταση. Και γι' αυτό ήθελα να σας αναφέρω ένα, μια πολύ μικρή φράση που το δείχνει αυτό εύγλωτα πιστεύω κάτι που είπε το 1912 ο αρχηγός της, ε, του πληθυσμού των Μπαχάη ε, στο Παρίσι πριν από, πάνω από 100 χρόνια. Όσο οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν έχουν πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε το μεγαλείο της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπες Κλάρος και τώρα δίνω το λόγο στα μέλη που μέχρι στιγμής έχουμε 7 αιτήσει για να λάβουν το λόγο. Θα κλείσω τώρα τον κατάλογο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και ζητώ από όλους τους ομιλητές να προσπαθήσουν να περιοριστούν σε δύο λεπτά. η κυρία Σταμπουλή καταρχήν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. President. Ε, η ελληνική νομοθεσία μέχρι το 2012 έχει ενσωματώσει ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών και απαγορεύουν κάθε διάκριση σε θέματα εργασίας και απασχόλησης ή και αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας και τις οδηγίες που προστατεύουν από σεξουαλική παρενόχληση και παρέχουν γονεϊκές άδειες. Οι οδηγίε αυτέ προστέθηκαν σε ένα ισχυρό πλέγμα προστασία τη μητρότητα που είχε διεκδικήσει και κερδίσει το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και μετά. Κατά την επταετία της κρίσης, η διεκδίκηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου δυσχεραίνεται από την υψηλή ανεργία και την υποστελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, αλλά και το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο βρίσκεται στο στόχαστρο των δανειστών. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ΕΡΣΤΑΤ, η γυναική ανεργία ήταν και παρέμεινε σημαντικά ψηλότερη από την ανδρική, η οποία όμως αυξήθηκε με γρηγορότερους ρυθμούς, μειώνοντας έτσι το χάσμα προς το χειρότερο. Αντίστοιχα, η μείωση του γενικού ποσοστού ανεργίας που παρατηρεί το 2015 ως το 2016 είναι ταχύτερη στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Όσο αφορά τα προγράμματα απασχόληση που εκπονούνται από το Υπουργείο Εργασία, γίνεται προσπάθεια να αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου ή και οικογενειακή κατάσταση. Στο πρόγραμμα για τη συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακή ζωή προσθέθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνική Αλληλεγγύη θέσει για παιδιά ανέργων μητέρων, ώστε έτσι να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασία. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη για τη στήριξη των αγροτησών σε συνδυασμό με την νομοθέτηση για του γυναικείου αγροτικού συνεταιρισμού που αφορούν την παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διακίνηση προϊόντων. Επίση, η Γενική Γραμματεία Ισότητα των Φύλων με ειδικά προγράμματα στηρίζει τη συμμετοχή των γυναικών σε τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών. Όσο αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, παρατηρείται σταθερή μικρή αύξηση ε, στην επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, όμως περίπου το μισό αυτής είναι επιχειρηματικότητα της ανάγκης. Η γυάλινη οροφή, όπως και το μισθολογικό χάσμα, παραμένουν και μένει να εκτιμηθεί η επίπτωσή του στο συνταξιοδοτικό χάσμα, με δεδομένο ότι το νέο ασφαλιστικό σύστημα, που είναι εν μέρει ανταποδοτικό σε σύνδεση με το εισόδημα, εφαρμόζεται από φέτος. Παραμένει επίσης εκτός κάθε υπολογισμού και αξιολόγηση η εργασία για το σπίτι και η φροντίδα για τα μέλη της οικογένειας. Η οικιακή εργασία και η φροντίδα που παρέχονται επαγγελματικά εξακολουθούν να είναι άλλοτε μη δηλούμενες και άλλοτε υποδηλούμενες, όπως έχουν τεκμηριώσει θαυμάσεις παρεμβάσεις της κυρία Κούνεβα. Και βέβαια ασκούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία από γυναίκες και ιδίω μετανάστρες. Η προσπάθεια των ελληνικών μηχανισμών που από πέρυσι επαναστελεχώνονται και στρέφονται και σε ελέγχους τέτοιων εργασιακών σχέσεων δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την οικονομική αυτονομία των γυναικών και να θεωρηθεί αυτή η αυτονομία ως ένας αναπτυξιακός πόρος σε όλες τις χώρες. Μπορώ να σας παρουσιάσω μερικά παραδείγματα από τη χώρα μου, τη Σλοβανία. Καταρχήν, πέρσι η κυβέρνηση της χώρας μου κήρυξε τη χρονιά αυτή ως χρονιά ε, του επιχειρήν για τις γυναίκες. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι σαφές από όλα αυτά, ότι υπάρχει μια πρόσθετη διάσταση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί με την εισαγωγή στον προπολογισμό συγκεκριμένων πρόνοιων ώστε τα εργαλεία του προπολογισμού να έχουν καλύτερη κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε λοιπόν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία με χρονικό ορίζοντα το 2020, αλλά το δίκτυο των γυναικών στη Σερβία που είναι ιδιαίτερα <clears throat> ενεργό έχει ε, ζητήσει από την κυβέρνηση και το δέχτηκε η κυβέρνηση κάθε χρόνο να υπάρχει μια έκθεση προς το Σερβικό Κοινοβούλιο σε σχέση με την πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται για τον νόμο αυτό εγγραφή στον προπολογισμό των μέτρων για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Είμαστε η πρώτη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που έχουμε χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο θετικό μέτρο και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε θεσπίσει μια στατιστική ανάλυση η οποία το υποστηρίζει. Προφανώ αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλέ γυναίκε στον κόσμο και σε πολλέ άλλε χώρε, <clears throat> ιδίω το θέμα τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη πρόσβαση εργαλείων για τι γυναίκε επιχειρηματίε και στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγε γυναίκε οι οποίε <clears throat> είναι ιδιοκτήτριε των επιχειρήσεων Ακολουθεί η κυρία Αριστίδου. Έχετε το λόγο. Στην περίπτωση της Κύπρου, το στρατηγικό σχέδιο για την ισότητα των φύλων καταγράφει τους ακόλουθους στόχους για την τόνωση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών. Καταπολέμηση της άνησης αμοιβή ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μείωση της ανεργίας και συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Περί τα τέλη του 2015, το Υπουργείο Εργασίας υλοποίησε συγχρηματοδοτούμενο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τίτλο «Δράσεις για μείωση του μισθολογικού χάσματος» που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010. Οι κύριες δράσεις που ελήφθησαν περιλαμβάνουν όπως την βελτίωση των μηχανισμών επιθεώρησης, τη δημιουργία εθνικού φορέα πιστοποίησης επιχειρήσεων, εξέταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τον εντοπισμό τυχών διακρίσεων στην αμοιβή, αλλά και άλλα ειδικά προσωρινά μέτρα όπως ήταν το πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, το κέντρο παραγωγικότητας Κύπρου που υλοποιεί προγράμματα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας όπως είχαμε και και το σχέδιο χορηγιών για ευέλικτες μορφέ απασχόλησης αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής ισότητας στο φύλλο στον εργασιακό χώρο. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, οι Κύπριες γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται πολλούς περιορισμούς που παρεμποδίζουν την οικονομική τους ενδυνάμωση. Θα πρέπει να προωθηθεί ο διαμοιρασμός ευθυνών ανάμεσα στα δύο φύλλα στο πεδίο του νοικοκυριού και της οικογένειας. Η επίτευξη της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών δεν είναι μια γρήγορη λύση, δεδομένου ότι απαιτείται η σφυριλάτηση δημοσίων πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση. Οι κοινοβουλευτικοί θεωρώ ότι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ο Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Ελ Γιασίρ για μία πτυχή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που είναι σημαντική για την υγεία των μητέρων είναι σημαντικό το να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, αναπαραγωγικής υγείας για τις γυναίκες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επανέλθει ο κανόνας ο οποίος εμποδίζει την χρηματοδότηση ε, ΜΚΟ που περιλαμβάνει υπηρεσίες άμβλωσης ή υποστήριξης της άμβλωσης. Αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχουν πιο πολλές μη θελημένες ε, ε, εγκυμοσύνης και επομένως <clears throat> πρόβλημα για την απασχόληση των γυναικών ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ερώτημα μου λοιπόν προς εσάς κυρία Γιασίν είναι βλέπετε τώρα να υπάρχει μια επίθεση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών γενικά και η εφαρμογή αυτού του λεγόμενου νόμου φήμωσης ε, κατά τον ΜΚΙΟ τι αποτέλεσμα θα έχει για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, την έγκαιρη επίτευξη των στόχων και τι επίπτωση θα έχει στην οικονομική ανάπτυξη και την χειραφέτηση των γυναικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούσλοβα ακολουθεί. Uh, from Ukraine. Από την Ουκρανία. Σούσλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποτελεσματική ισότητα στην Ουκρανία <clears throat> δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Υπάρχει ακόμα ένα χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας στην Ουκρανία. Αυτό ισχύει για το χάσμα το μισθολογικό, την πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης της επιχειρήσης <clears throat> και αυτό το χάσμα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα Είναι 30% αυτό το χάσμα στην Ουκρανία. Και ένας από τους λόγους για αυτή την στρέβλωση είναι η ανάπτυξη της, του διαχωρισμού σε επαγγέλματα. Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που θεωρούνται αποκλειστικά γυναικεία αποκλειστικά ανδρικά. Οι γυναίκες είναι οι πρώτες οι οποίες απολύονται και είναι δύσκολο να βρουν μια νέα θέση εργασίας. Περίπου 30% των αγγελιών για θέσεις εργασίας απαιτούν ο υποψήφιος να είναι άνδρας ή θα πρέπει <clears throat> να ε, εκπληρεί ορισμένες ε, απαιτήσεις σε σχέση με την ηλικία. Και στη συνέχεια οι υποψήφοι ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ερωτήματα για την υγεία τους και για συνέχεια υπάρχει πάντα το ερώτημα θα κάνετε παιδιά ή όχι. Υπάρχει ακόμα μια πτυχή που αναφέρθηκε επίσης σήμερα. Η νομοθεσία στην Ουκρανία εμποδίζει τις γυναίκες από το να ασχοληθούν με ορισμένα επαγγέλματα. Πάνω από 450 τέτοια επαγγέλματα αποκλείουν τις γυναίκες. Αυτό δεν είναι προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας, αυτό είναι μια διάκριση. Και υπάρχουν και διακρίσεις σε ό,τι αφορά την νυχτερινή εργασία των γυναικών, την εργασία κατά τη, διάτερα, <clears throat> διάρκεια διακοπών, όλα αυτά περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Θέλουμε λοιπόν κάποια από τα λεγόμενα προστατευτικά μέτρα να ακυρωθούν, να καταργηθούν, γιατί όλα αυτά οδηγούν σε αρνητικές διακρίσεις κατά των γυναικών και θέλουμε να ληφθεί υπόψη η απλήρωτη εργασία των γυναικών στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών. Πρέπει λοιπόν με αυτά τα μέτρα να αυξήσουμε συγχρόνως και τον αριθμό των γυναικών που είναι επιχειρηματίες. Η υποεπιτροπή μας για τα θέματα ισότητος εφέτος θα ασχολείται με τα εξή θέματα. Η ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές Επίσης, η χρήση, η ισότητα στις βιομηχανικές και πτωμιακές στρατηγικές ανάπτυξης. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε την κατάσταση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που είναι εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, άτομα που ανήκουν στην κοινότητα των Ρωμά, ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες προφανώς επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση και την ένοπλη σύραξη <clears throat> στην Ουκρανία. Οι ομάδες αυτές του πληθυσμού πολλές φορές υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και θέλω επίση να αναφέρω ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να επιτευχθούν αυτές οι λύσεις. Ευχαριστώ. Έχουμε μόνο 15 λεπτά για να κλείσουμε. Παρακαλώ στο τον πιο σύντομες οι παρεμβάσεις σας. Κυρία Μπιττική από το Κοσφοπέδιο. E, Καλημέρα σα και ευχαριστώ. Η δημοκρατία του Κοσφοπεδίου είναι νέα χώρα με πολλές προκλήσεις και στο θέμα της ισότητας των φίλων Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το ότι μιλούμε σήμερα για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών σήμερα. 11% είναι οι γυναίκες επιχειρηματίες με δραστηριοποίηση κυρίως στις υπηρεσίες με περιορισμένο ρυθμό εργαζομένων, ενώ τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως ανήκουν σε άντρες και δικούνται από άντρες. Η οικονομία μας είναι ακόμη στα σπάργανα, επιχειρηματι... επιχειρηματίες δεν υπάρχουν τόσο πολύ τους ή άλλους και οικονομική δραστηριότητα. Ε, δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως ο πόρος ε, αυτός, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητεί διαρκώς να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία. Παραμένει όμως ακόμη περιορισμένη αυτή. Η διαφθορά, η απουσία ανταγωνισμού, η απουσία πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένουν εμπόδια 8% ε, μόνο είναι το ποσοστό των γυναικών που κληρονομούν. Έχουμε λοιπόν εισαγάγει μια νέα διάταξη, νέο νομοθέτημα, που είχε σαν συνέπεια 620 οικογένειες κατά τη διάρκεια του 2014 να μπορούν να καταγράψουν συν ιδιοκτησία, συν ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε ακίνητο. Ένα μικρό βήμα, αλλά ε, σημαντικό πιστεύω. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την πρόσβαση στις επιχειρήσεις και στη διαχείριση της διοίκησης των επιχειρήσεων σε γυναίκες. παρουσία τους ξέρουμε ότι ωφελεί ιδιαίτερα και την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μια οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ματέρκη. Ε, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα-δύο σημεία. Η ενίσχυση της θέσης της γυναίκας ε, στην οικονομική ζωή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως. Για τα κορίτσια έχει τεράστια σημασία η εκπαίδευση, το δεκαετής πρέπει να είναι τουλάχιστον πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια. Έχουμε μπορέσει να αυξήσουμε από ε, ένα γύρο στο 15% στο 44% τα ποσοστά των γυναικών, των κοριτσιών που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Ταυτάχρονα και επιχειρηματίες ε, είναι πολλές ε, γυναίκες και ενισχύεται γενικά η απασχόληση των γυναικών. Για τα κορίτσια θα ξαναγυρίσω τώρα και υποστήριξη για την ε, εκπαίδευσή τους και πρόσθετη υποστήριξη οικονομική προς τις οικογένειες για να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο στις φτωχές οικογένειες ε, σε γυναίκες επί παραδείγματι άπορες ε, όταν πεθαίνει ο σύζυγός τους που καταβάλλεται ένα επίδομα επίσης γυναίκες που δουλεύουν στο σπίτι, σε σπίτια, ε, ε χωρίς να είναι δηλωμένη εργασία, τώρα καλύπτονται από την νομοθεσία. Είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται λοιπόν η οικιακή ε, εργασία. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα των γυναικών με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση ακινήτων ως εγγύησεων αλλά και κινητών ε, ως ενεχείρου για την εξασφάλιση δανείου από τις ε, τράπεζες. Επί παραδείγματι, μηχανήματα μιας επιχείρησης μπορούν να προσφερθούν ως ενέχειρο για την εξασφάλιση δανείου. Έχουμε συμπεριλάβει και στο Σύνταγμα ε, την, ε, το σύστημα των θετικών προτιμήσεων, ε, τα συστήματα της ευέλικτης εργασίας που ιδιαίτερα ευνοούν τις γυναίκες και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή της γυναίκας σε όλη την οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε. Τελευταία ομιλήτρια κυρία Γιούνες από την Τινησία. Ευχαριστώ η Μισελία Τούνες από το Κοινοβούλιο της Τινησίας. Ήθελα να σας μιλήσω για ένα πρόβλημα όλων των γυναικών, πιστεύω. Η Τινησία είναι μια μικροσκοπική χώρα στην ε, Βόρεια Αφρική που πάντοτε τη στήριζε η δύναμη των γυναικών της. Πάντοτε οι γυναίκες εργάζονταν σκληρά και έδιναν πολλά στη χώρα. Πάνω από 50 χρόνια ε, ε, είναι το διάστημα που κοιτάζουμε την νομοθεσία, την νομοθεσία που μπορεί να ενθαρρύνει τις γυναίκες. Και παρόλα αυτά, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες κατέχουν όλα τους τα νόμιμα δικαιώματα στην Τινησία. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ε, δεν είναι πλήρης. Εγώ λοιπόν ως βουλευτής θεωρώ ότι υπάρχει χάσμα. Χάσμα μεταξύ του τι λέει ο νόμος και το τι γίνεται στην πράξη. Πώς εφαρμόζεται ο νόμος. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς να πιέσουμε οι νόμοι να ε, τηρούνται, ώστε οι γυναίκες να έχουν στα χέρια τους όλα τους τα δικαιώματα. Δικαίωμα στην οικονομία, την οικονομική παραγωγή, την εκπαίδευση, την υγεία, σε όλα για να έχουμε μια κοινωνία ισορροπημένη, μια κοινωνία χειραφατημένη, για να το πω. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που βλέπω να επαναλαμβάνεται στη χώρα μου. Η γεωργία βασίζεται στις γυναίκες. Οι γυναίκες δουλεύουν στα χωράφια. Ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο προσφάτως, πάνω από ένα χρόνο τώρα, ένα νόμο για την ισότητα των ανιδών, των μισθών. Ένα νόμο για την κοινωνική ασφάλιση. Διότι πρόκειται για δουλειά με μισθό κάποιες φορές τουλάχιστον ε, τον μισό του αντίστοιχου αντρικού και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Και ως σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν τηρείται αυτός ο νόμος. Πώς λοιπόν μπορούμε στην πράξη, στην καθημερινότητα να επιβάλλουμε την τήρηση του νόμου, πώς να επιβάλλουμε την τήρηση του νόμου, διότι αυτοί οι νόμοι θα επιτρέψουν να αλλάξουν οι τροπίες και φτάνω και στο συμπέρασμά μου ότι με τους νόμους χρειάζεται αλλαγή στις νοτροπίες. Εκεί πιστεύω είναι η ουσία του προβλήματος. Καλοί οι νόμοι πρέπει να υπάρχουν, ωραία είναι τα κοινοβούλια και η πολιτική το δικό μα κοινοβούλιο με 30% γυναίκε, σε επίπεδο ε, ε ανώτατη εκπαίδευση και πτυχιούχων 65% τουλάχιστον είμαστε γυναίκε, αλλά σε επίπεδο νοοτροπία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλου για τι παρεμβάσει του. Δεν υπήρξε καμία ισορροπία στα φύλλα που πήραν το λόγο. Έτσι είναι η ζωή. Τώρα ο λόγος πάλι στους συμμετέχοντες στο πάνελ. Θα σας παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ σύντομοι, διότι έχουμε μόνο 5 λεπτά. Κυρία Ελ Γιασίρ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα σχόλια και όλα τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Απλώ να σα πω ότι είναι πραγματικά ανθαρρυντικό να ακούσουμε από τόσο πολλού από εσά ότι υπάρχει υποστήριξη για την ιδέα που τονίστηκε σήμερα σε αυτό το εργαστήριο ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη εγγραφή στον προϋπολογισμό για τα θέματα ισότητος, να ξεπεράσουμε τους ε, διακριτικούς νόμους και τις πρόνοιες. Επομένως, αυτό το υποστηρίζω. Και δύο ακόμα πρόσθετα σχόλια. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αναφέρθηκε από την ε, Ελληνίδα βουλευτή για τις προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ισότητας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτό ακριβώς ε, αναφέρουμε τώρα όταν δεν εναπόκειται μονάχα σε μια χώρα, είναι κάτι που αφορά όλε τι χώρε. Όταν πρέπει να ξανασκεφτούμε τι μακροοικονομικέ πολιτικέ, όχι μονάχα σε μια χώρα που παίρνει βοήθεια, αλλά και σε ό,τι αφορά του φορεί που δίνουν αυτή τη βοήθεια. Αυτέ είναι οι αλλαγέ οι οποίε συμβαίνουν και τώρα ακόμα και το Δούνου του αρχίζει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά γιατί αναγνωρίζουν ότι αυξάνονται οι ανισότητε μέσα από τις πολιτικές που ισχύουν. Επομένως χρειάζεται μια συμβολική συνολική προσπάθεια. Και τέλος, για ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, για την πρόσβαση στην ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι γενικότερο και το έχει θίξει και ο συναδελφός μου η ισότητα των φύλων έχει και οικονομικό όφελος και οι στατιστικές που σας έδωσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από το γεγονός αυτό. Υποστηρίζουμε την οικονομική την ισότητα των φύλων για να έχουμε και οικονομικά ωφέλη, αλλά καταρχήν αυτό είναι ένα δικαίωμα και πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο δικαιωμάτων. Είναι κανονιστικά πλαίσια τα οποία έχουμε πραγματικά την συλλογική ευθύνη να τα υποστηρίξουμε. Ακόμα και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν λοιπόν υπήρξε υποχώρηση ή παναχώρηση, δυστυχώ τα πράγματα σε ορισμένε φορές πηγαίνουν προς τα πίσω. Υπάρχουν πολλοί υποστηρικτέ των δικαιωμάτων ισότητος, είτε στην κυβέρνηση είτε στην κοινωνία των πολιτών, <clears throat> ότι τώρα αντί να υπάρξει πρόοδος, ο αγώνας του είναι μοναχά να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα και πάντα θα πρέπει να προσεκτικοί σε σχέση με τις διατυπώσεις μας. <coughs> Μπορούμε να μιλάμε για οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά πότε δεν θα το κάνουμε αυτό σε βάρος των δικαιωμάτων και των κανονιστικών πλαισίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Κλάρος. Ξέρετε ότι υπάρχει μια απέραντη φιλολογία και σύνολο μελετών για τη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ευμάρειας αφενός και των περιορισμών που ασκούνται στις γυναίκες και ιδίως στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και τα δικαιώματά τους. Δεν έχω το χρόνο τώρα να τα διεξέλθω όλα αυτά. Σας δώσω μόνο δύο-τρία παραδείγματα. Ξέρουμε ότι παραδείγματο χάρη όταν πάμε σε έναν κόσμο που έχει χαμηλότερη διαφορά ανδρών και γυναικών σε απασχόληση, αυτό αλλάζει και την ισορροπία εξουσία μέσα στην οικογένεια. Όταν οι γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα, γιατί εργάζονται και γιατί είναι μορφωμένες, έχουν μεγαλύτερη επιρροή μέσα στο σπίτι και τώρα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των οικιακών πόρων, περισσότερε ευκαιρίε για επένδυση, καλύτερη βοήθεια των παιδιών, επομένως τίθενται οι σπόροι για την επόμενη γενιά η οποία θα είναι πιο ε, ανεπτυγμένη σε ανθρώπινο επίπεδο. Όταν λέμε ότι η ισότητα των φύλων είναι καλή σε επίπεδο οικονομικό, αυτό δεν είναι μια δογματική δήλωση που έχουμε διατυπώσει, είναι πραγματικότητα γιατί υπάρχουν βαθιές ρίζες στην οικονομική, στις οικονομικές πολιτικές αυτού του φαινομένου και είναι και η εμπειρία των χωρών μας. Τέλος, επειδή δεν έχω χρόνο, να αντιμετωπίσω το σχόλιο που έγινε από την εκπρόσωπο της Ουκρανίας όταν είπα ότι στην Ουκρανία όπως και στη Ρωσία υπάρχουν πολλαπλές ε, μορφές περιορισμού για την πρόσβαση σε επαγγέλματα. Η δική μου εμπειρία με συναντήσεις με αξιωματούχους αυτής της χώρας είναι ότι υπάρχει μια πολλές φορές <clears throat> πατερναλιστική αντιμετώπιση οι οποίοι θέτουν περιορισμούς υποτίθεται για την προστασία των γυναικών αλλά σας λέω με ποιο τρόπο οι γυναίκες οδηγοί του μετρό της Μόσχας προστατεύονται από τέτοιους περιορισμούς. Είναι, είναι τόσο επικίνδυνο να οδηγεί κανείς τους σειρμούς του μετρού, του μετρό στη Ρωσία. Όχι. Πολλές φορές αυτοί οι περιορισμοί είναι ιστορικού χαρακτήρα, υπάρχουν στην νομοθεσία μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, εξακολουθούν να γίνονται. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την έλλειψη πολιτική συναφέτησης των γυναικών. Οι άνδρες κάνουν του κανόνε, οι άνδρες περνάνε αυτές τους ανόητες μορφές νομοθεσίας και αυτές οι αλλαγές θα γίνουν όταν οι γυναίκες έχουν την πολιτική εξουσία και έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινοβούλια όταν ανέλθει από το 20% που είναι αυτή τη στιγμή σε κάτι πλησιέστερο από τα 50% ίσως στο, στο μακρινότερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος της ε, συνόδου αυτής. Εν συμπεράσματι <clears throat> να σας πω ότι υπάρχουν δύο βασικές ιδέες οι οποίες προήλθαν από τις διάφορες παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς την ισότητα των φύλων και δεν θα υπάρξει ισότητα των φύλων χωρίς την οικονομική χειραφήτηση των γυναικών γιατί όπως λέγεται πολλές φορές η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι ένας κέριος μοχλός για να υπάρξει περιεκτική ανάπτυξη σε οικονομικό επίπεδο και επομένως βιώσιμη ανάπτυξη. Και η δεύτερη ιδέα, εμείς οι νομοθέτες μπορούμε να παίξουμε ένα κέριο δρόμο στο να διαμορφώσουμε και να ακυρώσουμε νόμους οι οποίοι έχουν διακριτικό, διακριτικό χαρακτήρα και μπορούμε να επιτύχουμε με την νομοθεσία να βελτιώσουμε την πραγματικότητα και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε εδώ. Να σας υπενθυμίσω ότι τώρα είμαστε όλοι καλεσμένοι στο εστιατόριο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έχει ξεκινήσει πριν από ένα λεπτό η τελετή μας για το βραβείο ίσως Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και ευχαριστώ τους ομιλητές μας, εισηγητές. Θα τα πούμε στο σχέδιο των